Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Λοιπόν, έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις Οπότε γκρίνονται και τα πρακτικά. Το ΕΛΚ έχει ζητήσει τους εξής διορισμούς. Τζοβάνι Λαβία στη θέση της κυρίας Σατόρη για την αντιπροσωπεία με τη σχέση των χωρών των Άνδεων και την αντιπροσωπεία Ευρώπης Λατινικής Αμερικής. Η κυρία Σατόρη, μέλος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη ΣΥΠΑ, Φαμπρίτσιο Γκαρτών, μέλος αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Ινδία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι, οπότε εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας με διάρκεια ε, μιας ώρας. Ξεκινάμε με το θέμα κράτος δικαίου στη Ρωσία. Έχουμε η κυρία Γιάκονσάρη, την κυρία Γιάκονσάρη θα λάβει πρώτη τον λόγο ως συντάκτρια των ψηφισμάτων. Για 1,5 λεπτό. Πού είναι η κυρία Γιάκονσάρη? Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία είναι τέρι. και στενοί συνεργάτες σε κάποια πράγματα. Θα έλεγα και φίλοι. Και οι φίλοι μπορεί να είναι ανοιχτοί, μπορεί να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Και αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, καλά κάνουμε που αγχωνόμαστε και ανησυχούμε για τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία. Αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία των πολιτών, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διότι ε, υιοθετείται κάποιο νομοθέτημα που τα επηρεάζει όλα αυτά. Ε, είναι εκπληκτικό το ότι οι οργανώσεις όπως Friedrich Herbert και Conrad Adenauer που είναι οργανισμοί με διεθνή φήμη στον τομέα της οικοδόμησης δημοκρατίας και δημοκρατικών θεσμών οι οργανισμοί αυτοί ε, είναι θύματα αυθαίρετων μέτρων και υποφέρουν στα χέρια των αρχών. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το θέμα του νόμου για τους ξένους ε, ε, πράκτορες κατά κάποιο τρόπο που εφαρμόζεται αυτός ο νόμος στα μέλη αυτών των οργανισμών. Και αυτό υπολείπεται των ε, διεθνών προδιαγραφών. Είναι κάτι που το καταδικάζουμε. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τεθούν αυτά. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε ενδελεχώς τα ζητήματα. και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δεχτεί αυτά που λένε οι Υπουργοί Εξωτερικών για τη Ρωσία. Σα ευχαριστώ κυρία Γιακονσάρη. Η κυρία Κορνέλισεν για μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά το να την κατηγορούμε ότι έχει και κατασκόπους υποστηρίζοντας τις ε, ρώσικες ΜΚΟ δεν μας φέρνει πιο κοντά. Ε, το ύφο διακυβέρνηση του κυρίου Πουτίν είναι η καταστολή των ΜΚΟ, των ε, ακτιβιστών και των μειονοτήτων. Ούτε μία σχέση δεν έχει με εξυγχρονισμό και σταθερότητα και μπορεί να οδηγήσει μόνο σε περισσότερη απομόνωση της Ρωσίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ταξίδι ε, με απαλλαγή θεώρησης ε, για τους Ρώσους αξιωματούχους όσο δεν απαγορεύεται η βίζα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του κυρίου και Από την άλλη ε, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει γρήγορα, να δίνει γρήγορα βίζα σε Ρώσους που υποφέρουν από πολιτικές διώξεις για να μην έχουμε άλλες αυτοκτονίες και απαγωγές. Μετά, οι νόμοι που πέρασαν αυτή την εβδομάδα στην Δούμα κατά της ε, ομοφιλόφιλης προπαγάνδας, όπως λέγεται, και για την προστασία των ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων. Άλλη μία υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσία παραβιάζουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργούν ε, έδαφος για πολιτικές διώξεις και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ και αντιβαίνουν τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διάλογο για τη βίζα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγαλών το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κορνέλισεν κυρία Ούχιλαντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά λόγια για το απλήγματα που δέχεται δημοκρατία στη Ρωσία. Τα είπε η Δύση. Σε πολλέ συνόδου κορυφή υπόθηκαν αυτά. Ψηφίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πολλά σχετικά ψηφίσματα. Και μάλιστα τελευταία τετραετία. Αποτέλεσμα, τίποτα, καμία αλλαγή. Τώρα όμως ήρθε η ώρα η Ευρώπη να κινηθεί. Και να αντιδράσει έναντι αυτών που βλέπουμε να συμβαίνουν στη Ρωσία. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό όταν είχαν οι πιέσει τη δημοκρατία στη ρωσική δημοκρατία και θα πρέπει να ε, κινηθούμε κατά του νόμου Μαγνίσκη. Και η κοινωνία των πολιτών σε όλη τη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί. Θα πρέπει η Επιτροπή του Ελσίνκη εντός της Δύσος να ανασυσταθεί για να υποστηρίξει την πολιτική αντιπολίτευση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών που μάχεται για τα δημοκρατικά της δικαιώματα και τα συνταγματικά της δικαιώματα στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγκάλσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κυρία Κορνέλισεν επεσήμανε πως ε, η Ρωσία είναι, λέει, στρατηγικός τέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται αυτό σε επίσημα έγγραφα. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ε, το εάν θέλουμε να διατηρηθεί κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο να φανταστούμε το πως ένα στρατηγικός εταίρος που κρύβει τον φόνο του Μαγνίτσκι δεν επιτρέπει στην ανεξάρτητη επιτρέπει την λειτουργία της δικαιοσύνη, ε, τον ΜΚΟ, διώκει ανθρώπους όπως τον Χόντορκόφσκι. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία σαφώς επιδεινώνεται. Οι εκλογές είναι στιμένες και αντιδημοκρατικές. Οπότε θα θεωρούμε πως είναι στρατηγικός εταίρος αυτή η χώρα. Ε, αν πιστεύουμε στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ρωτηθούμε. Ευχαριστώ. Μπερζιά για δύο λεπτά. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το Σοβιετικό μπλοκ και μετά η Ρωσία δυσκολεύεται να βρει το δρόμο της δημοκρατίας με σκαμπανεβάσματα. Με το που πήγε στο Κρεμλίνο ο Πούτιν ε, δρομούμε αντί να προοδεύουμε. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα μας αφήνουν άναυδους. Μπορεί κανείς ε, να αναρωτηθεί για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, γιατί η υπόθεση Μαγνίτσκι είναι ένα μόνο παράδειγμα μεταξύ άλλων. Και ε, δεν έχω μόνο αμφιβολίες έχω κάτι ισχυρότερο. Εγώ δεν έχω προσωπικά μία αμφιβολία. Ε, ε, η Transparency International μας δίνει τα σχετικά αποτελέσματα και δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Και στην 189η θέση βάση της Amnesty International. Είναι ένα κατασταλτικό παζλ το κυβερνητικό σχήμα στη Ρωσία. Πρέπει να καταχωρηθούν όλοι οργανισμοί ε, στο μητρό των αλλοδαπών, έτσι ονομάζεται, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Ενώ πρόκειται για μη κυβερνητικέ οργανώσει και είδαμε και τι συνέβη στι τελευταίες εκλογές. Η φρασιολογία που χρησιμοποιείται μας θυμίζει εποχές Στάλιν. Ε, ε, το βραβείο ε, Ζαχάροφ ε, είναι ένα από τα θύματα του καθεστώτος και ας χαιρετήσουμε το θάρρος και το κουράγιο των αντιφρονούντων. Ο απολυταρχισμός της Ρωσίας και ο νεοφιλελευθερισμός χωρίς κανένα όριο συνδυάζονται σε ένα εκρηκτικό μίξ. Ποιο μπορεί να είναι ο, ο δημοκρατικός απολογισμός, ο απολογισμό σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί έχουμε εταιρική σχέση με ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με τη Ρωσική Ομοσπονδία για αυτό το θέμα. Σε τι χρησιμεύει ακριβώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Βέρζια. Λίσεκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, Επίτροπε. Περίπου 150 μέλη έχουν υπογράψει για να δημιουργηθεί ένα για την ανάθεση του, του, του βραβείου Ζαχάροφ για ένα μνημείο, για να αποδοθεί το μνημείο Ζαχάροφ να δοθεί σε μια οργάνωση που είναι μια οργάνωση με μέλη τα οποία δέχονται αρνητική αντιμετώπιση από τις ρωσικές αρχές. Τα πολιτικά κόμματα, οι προσφυστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι όλοι διώκονται. Πρέπει να απευθυνθούμε στην ύπατη εκπρόσωπο, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον πρόεδρο του Συμβουλίου, να κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να ξεκινήσουν συζητήσεις με τη Ρωσία σε όλα τα επίπεδα, για να πιστήσουμε την προσοχή στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, διότι δεν υπάρχουν πλέον στη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίσεκ. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι εισηγητέ. Περνάμε στου ομιλητέ των ομάδων. Κύριο Πόσολτ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μία συνάδελφο μίλησε για Ρώσους συναδέλφους ε, και Ρώσους φίλους. Οι δικοί μου οι Ρώσοι φίλοι δεν είναι στο καθεστώς Πούτιν. Είναι είτε νεκροί όπως ο Μαγνίτσκι, όπως η κυρία Εστιμέροβα, η κυρία για με την οποία είχα στενή συνεργασία, ή είναι κάπου στη Σιβηρία και σπάνε πέτρες όπως ο κύριος ε, Χοντορκόφσκι ή ο κύριος ε, Λέμπεντεφ ή ο κύριος Ναβάνη. Στραγγαλίζονται όπως το Memorial και άλλοι οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Αντενάουερ και Έμπερτ ή φυλακίζονται όπως οι γυναίκες των Πούσιράιωτ ε, που επίσης θα ήθελα να αναφέρω. Και αυτό ξεκαθαρίζει πως έχουμε να κάνουμε με ένα στιγνό καθεστώς και θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα, όχι να μην μιλάμε για λόγους πρώτων υλών. Σε αυτήν την κοινότητα υπάρχουν και κοινέ αξίες και ποινέ βάσει. Γι' αυτό πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα στη Ρωσία. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Κύριε Μουνίθ. Ανησυχούμε και εμείς για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία, κυρίως σε σχέση με τον χαρακτηρισμό ως ξένων πρακτόρων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, το πώς μεταχειρίζεται η κυβέρνηση την αντιπολίτευση, υπόθεση Μαγνιέτσκι και άλλες, η προπαγάνδα σε σχέση με την ομοφιλοφιλία. Δεν πιστεύουμε όμως ότι ε, τα επαναλαμβανόμενα κατεπήγοντα ψηφίσματα για την ε, Ρωσία χρησιμεύουν σε κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ε, πρέπει να ε, παγιωθεί ο πολιτικός διάλογος, να χρησιμοποιήσουμε τις συνόδους κορυφής για να εγείρουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και μην ξεχνάμε ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ε, πολλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται την ίδια μεταχείριση. Ποιο είναι το νόημα των επαναλαμβανωμένων ψηφισμάτων? Ευχαριστούμε, αγαπητοί συνάδελφε. Τάκουλα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι σε θέση να πω μερικά λόγια σήμερα για το κράτος δικαίου στη Ρωσία. Ανησυχώ για αυτά που συμβαίνουν. Και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος διότι μια φιλανδική αντιπροσωπεία είναι εδώ και παρακολουθεί τη συζήτηση. Ε, και, αυτή, και η Φιλανδία γνωρίζει πολλά για τη Ρωσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κόσμος στη Ρωσία, ανεξάρτητα τις θεσμικές του πεπιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ, πρέπει να απολαμβάνει πλήρως των πολιτικών του δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες έχουμε εμπορικέ σχέσεις, ότι οι χώρες αυτές σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την πραγματική έννοια του όρου. Η Ρωσία είναι ένας σημαντικός εταίρος δεν θα πρέπει λοιπόν να εθελοτυφλούμε όσον αφορά ε, τι πράξει τη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει σαφέστατο μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που να γίνονται σεβαστά. Σα ευχαριστώ. Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ήμουν ένας από αυτούς που ήθελε η Memorial, η οργάνωση αυτή, να λάβει, να παραλάβει να... το βραβείο Ειρηνη Νόμπελ, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Υπάρχουν δύο Ρωσίες. Έχουμε την επίσημη Ρωσία από τη μια μεριά, το κράτος. Και έχουμε αυτή τη Ρωσία λοιπόν που πιστεύει στη χρήση δύναμης που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απ' την άλλη έχουμε την άλλη Ρωσία η άλλη Ρωσία δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι αδύναμη. Είναι αδύναμη. Εν μέρη λόγω της αδράνειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της ανικανότητάς της. Ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταδικάζουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε, στις χώρες Χ, Ψ και Ω αλλά δεν κατακρίνουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την Κίνα γιατί έχουμε πολύ μεγάλο όγκο εμπορικών συναλλαγών με αυτές. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό Κύριο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη Ρωσία. Η ρωσική κυβέρνηση είναι ένα γκαγκστερικό καθεστώς και εξάγει το κράτος της αδικίας στην Δύση και εντωμεταξύ οι δυτικές κυβερνήσεις ακολουθούν μια πολιτική κατευνασμού. Το 2006 πράκτορες του ρωσικού κράτους ε, δολοφόνησαν τον ε, ψηφοφόρο μου, τον κύριο Λιτβινέγκο, σε μια πράξη κρατικής τρομοκρατίας. Ο Ντέιβιτ Κάμερον δεν ε, τήρησε την υπόσχεσή του για να αποκαλύψει το τι συνέβη. Ανταυτού κατέληξε συμφωνία με τον πρόεδρο Πούτιν. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν θα αφήσει να βγουν σημαντικά στοιχεία στην δίκη ε, που αποδεικνύουν ε, τη συμμετοχή του ρωσικού κράτους. Δολοφονούνται από το ρωσικό κράτος άνθρωποι στους δρόμους του Λονδίνου και η Βρετανική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Οποιαδήποτε συνεργασία με τη Ρωσία σε ζητήματα νομικά και ασφαλείας πρέπει να αποκλειστεί μέχρι να υπάρξει πραγματικό κράτος δικαίου. Σας ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι ομιλητές από πλευράς ε, των ομάδων. Περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Πρέντα. Πρόεδρε, η κυρία Μούνης είπε πριν από λίγο πως ε, δεν είναι πολύ καλή ιδέα να συζητάμε το θέμα της Ρωσίας ε, την Πέμπτη το απόγευμα και κυρίως όχι επί ευκαιρία ενός ψηφίσματος. Δεν είμαι σίγουρος ε, πως ε, μια συζήτηση για τη Σύνοδο ΕΕ Ρωσίας θα ήταν καλύτερη ιδέα. Έχουμε Δεν έχουμε κατορθώσει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής για την Ρωσική Ομοσπονδία. Οι μη κερδοσκοπικέ οργανώσεις ε, στη Ρωσία έχουν δεχθεί εκφοβισμό λόγω της, ε, του νέου νόμου που εγκρίθηκε στη Δούμα το Νοέμβριο του 2012. Υπάρχει κράτος δικαίου άραγε στη Ρωσία. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα για ένα λεπτό ο κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χτες μιλήσαμε εδώ πέρα για την ανάγκη συνέπειας της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και σήμερα κατονομάζουμε τη Ρωσία. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε τη χειρότερη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά την ε, Σοβιετική εποχή και σήμερα ζητάμε την ανάκληση του νόμου περί ξένων πρακτόρων καθώς προσπαθεί να ε, χαρακτηρίσει την οργάνωση Memorial και άλλες ως πράκτορες και προδότες και πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τον διάλογο με την ε, ρώσικη κοινωνία των πολιτών. Μήπως θα παρακολουθούμε ενώ αυτή εξαφανίζεται. Επίσης ε, δεν... υπάρχει ένας νέος νόμος ο οποίος ε, απαγορεύει την πληροφόρηση για τη μη παραδοσιακή σεξουαλικότητα. Οι δε τρεις φόνοι που έγιναν ε, στη Ρωσία τον Μάιο αποδεικνύουν πως το δικαίωμα αυτό βρίσκεται υπό απειλή. Σας ευχαριστώ. Σόνικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι μια χώρα που μας έδωσε τον Τζενίτιν, τον Ζαχάροφ, αλλά και τον Στάλιν και τους Μπολσεβίκους. δεν μπορεί να προσέξει τους και να φροντίσει τους πολίτες της. Το κράτος δημιουργεί τους δικούς του μηχανισμούς. Το κράτος δεν μπορεί να απαλλαγεί από το σταλινισμό, από το φορτίο του σταλινισμού. Το κράτος φοβάται τους ελεύθερους πολίτες. Ο Σολτζενίτσιν, ο Ζαχάροφ ήταν πηγή περηφάνειας για τη Ρωσία οι ακτιβιστές της Memorial και οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι είναι σήμερα εκείνοι που είναι η υπερηφάνεια της Ρωσίας. Το κράτος προσπαθεί να τους υπονομεύσει και να τους κατονομάσει σαν προδότες και σαν ξένους πράκτορες. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Ρωσία να ξεπεράσει τα συμπλέγματά της. Θα πρέπει να πούμε «Ρωσία, είσαι υπέροχη χώρα». Αλλά για να γίνει μεγάλη δεν πρέπει να καταστρέφει την αντιπολίτευση και τον ελεύθερο Και κλείνω. Πρόεδρε, δεν, δεν πρέπει λέω να διώκει Ρωσία το λαό σου. Ο κ. Σαντσμπέρκης έχει κάποια ερώτηση να θέσει στον κύριο Σόνικ. Μια παρατήρηση, παρατήρηση. Πρόεδρε, αν θέλουμε διάλογο με τη Ρωσία, πρώτο βήμα θα είναι να διορθώσουμε τον τίτλο. Κύριε Λαντσμπέργκης, έχουμε τη διαδικασία και HDI και έχουμε μπλε κάρτα. Μπλε κάρτα σημαίνει ερώτηση στον ομιλητή. Ε, μάλλον θα σας βάλω στον κατάλογο των ομιλητών για το HDI. Α, ερώτηση στον κύριο Σόνικ, εντάξει. Μία ερώτηση λοιπόν. Εάν θεωρεί πως ε, πρέπει να διορθωθεί ο τίτλος ε, της έκθεσης από το κράτος δικαίου στο κράτος ε, Κρεμλίνου ή κάτι ανάλογο. Ευχαριστώ. Κύριε Σόνικ. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον κύριο Λαντσπέρκης. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι πιο ε, στεναρός. Μας δίνει όμως τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία και έτσι έχω αρκετούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να μιλήσουν όλοι, αλλά πρέπει να είμαστε κάπως πιο αυστηροί. Λοιπόν, η κυρία Σαγιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση για το κράτος δικαίου η Ρωσία είναι πραγματικά απαραίτητη, διότι είναι στρατηγικός εταίρος της Ένωση η Ρωσία και άρα πρέπει να γύρουμε αυτά τα ζητήματα για να υπεραμεινθούμε των δημοκρατικών αξιών είτε στην Ευρώπη είτε ε, στην επικράτεια των στρατηγικών μας εταίρων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Η Ρωσία άρχισε να χαρακτηρίζει τις μη κάπα ως ξένους πράκτορες. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, πρέπει να καταχωρηθούν σε ένα αντίστοιχο μητρό και σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ένα μεγάλο πρόστιμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ευελπιστώ να τεθεί στο ε, δυνατό επίπεδο. Δεν θα ακούσουμε κάποιον άλλον στην ε, διαδικασία και Έκλεισε ο κατάλογος. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Ρουέδα. Ευχαριστώ. Η κατάσταση στη Ρωσία πραγματικά είναι συμπτωματική των συνολικών προβλημάτων σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαρακτηρίζεται από ένα ασφικτικό δικαίωμα που προσπαθεί να περιορίσει τα δικαιώματα της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι πως υπάρχει ομοσπονδιακή νομοσπονδία για την ομοφιλόφιλη προπαγάνδα που θα αυξήσει την ε, βία και τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ. Αλλά επίσης οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για να σταματήσει αυτή η ε, νομοθεσία για την λεγόμενη προπαγάνδα. Γι' αυτό θα ήθελα στο κείμενο που θα ψηφίσουμε να μπει ένα συγκεκριμένο αίτημα για να ζητήσουμε από την Δούμα να σταματήσει η συζήτηση για τέτοιους νόμους. Δεν έχει γίνει, αλλά ε, νομίζω πως και το θέμα της νοοτροπίας είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ρωμέβα. Ε, και ακολουθεί. Ευχαριστώ. Συζητούμε για το κράτος δικαίου στη Ρωσία και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη 10η Απριλίου 2010 όταν ο πρόεδρος Λεκατσίνσκι πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας σκοτώθηκε και παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα η Ρωσία αρνείται να παραδώσει το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Αυτό παρεμποδίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις έρευνες των πολωνικών αρχών. Οι ρωσικές αρχές είχαν χρόνο στη διάθεσή τους για να διεξάγουν τη δική τους έρευνα. Τον αρνούνται τώρα να παραδώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σίγουρα δεν ευθυγραμμίζουν με βασικές αξίες του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστούμε για Σοβιέτσκα τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τους περασμένους μήνες Βιώσαμε γίναν μάρτυρες μάλλον μιας καταστολή ε, από πλευρά των ρωσικών αρχών. Δυστυχώ ε, οι διερμηνεί αδυνατούν να παρακολουθήσουν ε, μια τέτοια ταχύτητα. Είναι λοιπόν <coughs> πάρα πολύ ανησυχητική κατάσταση στη Ρωσία. Ακούμε ε, επανειλημμένα ότι είναι απολυταρχικό κράτος η Ρωσία και ότι δεν υπάρχει ούτε ελευθερία ούτε ανεξαρτησία. Οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική της για τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε το, την ουτοπία ε, μιας εξυγχρονισμένης Ρωσίας, ε, διότι δεν κάνει τα δέοντα το Κρεμλίνο. Εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και θα αφήσουμε τα κράτη-μέλη να συνομιλούν με τις δροσικές αρχές. Ευχαριστούμε, Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για τη Ρωσία λοιπόν. Αναμφισβήτητα πολλοί αρχίζουν να έχουν υποψίες, να πιστεύουν τα πράγματα δεν είναι όπως θα έπρεπε στη Ρωσία και κυρίως όσον αφορά τον Πούτιν και τους συναδέλφους του Πούτιν δεν έχουν μεγάλο σεβασμό για τα πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών τους και δεν έχει νόημα να διαβάζουν περισσότερα για αυτά που συμβαίνουν εκεί. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρή και πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας μαζί τους και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ελευθερία των πολιτών και τα πολιτικά τους δικαιώματα και ανοιχτέ και διαφανείς συνομιλίες πρέπει να λάβουν χώρα και θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα ηθικά πρότυπα, τα κοινά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κόρολα. Ευχαριστώ. Ως ε, μέλος ε, του ΟΑΣΕ και ως χώρα που έχει υπογράψει πολλές συμβάσεις του η Ρωσία πρέπει να σέβεται τους, τις αρχές του κράτους δικαίου. Οι πρόσφατες δίκες στη Ρωσία ήταν ηχητικές. Αναφέρθηκε ο Μαγνίτσκι, ο Χοντορκόφσκι και η κυρία Πολιτκόφσκαγια στο ψήφισμα, αλλά πρόκειται απλά για λίγα τρανταχτά παραδείγματα με τα οποία η Ρωσία αψηφά βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Η κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία υποφέρει το, η ιδέα αντιμετώπιση των ομοφυλόφιλων είναι διακριτική, πραγματικά είναι διάκριση. Η Ρωσία είναι σημαντικός ε, εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τα πει αυτά η κυρία Άστον. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και η κυρία Φοντούν und Hohenstein. Mm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι συζητάμε αυτό το ψήφισμα και για το ότι αναφέρεται σε ΜΚΟ, γιατί χωρίς ΜΚΟ δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι οργανωμένη. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εργάζονται διεθνώς για την ειρήνη, μοιραία, ε, χρηματοδοτούνται από άλλες χώρες, το ίδιο και το Memorial. Ε, λογικό είναι να παίρνουν λεφτά από το εξωτερικό, αλλά το να τους λέμε πράκτορες είναι χιδέα συκοφαντία και προσβολή προς τη δημοκρατία και στις αρχές ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών. Ο Στάλιν πίστευε στο ότι αν πεις ένα ψέμα 100 φορές γίνεται αλήθεια. Και ο Γκέμπελς το ίδιο είχε πει και να είμαστε πάλι εδώ. Βλέπουμε α, ε, χιδέα ψέματα σε μια χιδέα κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Και εδώ πέρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο κύριος Λεβαντόφσκι θα μιλήσει τώρα εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτή η συζήτηση δείχνουν τι αυξανόμενε ανησυχίες τη Ευρωπαϊκή Ενώση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό αφορά τη γενική κατάσταση αλλά και ξεχωριστές περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σήμερα. Αυτό είναι κάτι που εθίγει επανειλημμένος από την ύπατη εκπρόσωπο, την Κάθριν Άστον. Ναι, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξαμε μάρτυρες επιδίνωσης του πλαισίου αντός του οποίου η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί στη Ρωσία. Πιο συγκεκριμένα αυτό γίνεται μέσω νέων νόμων με ιονή νόμιμο τρόπο. Κοινό στόχο των νόμων για την προδοσία, για τους ξένους πράκτορες, για τις διαδηλώσεις και πιο πρόσφατα για την ομοφιλοφιλική προπαγάνδα φαίνεται να χρησιμοποιεί να περιορίζουν το χώρο για ανεξάρτητη κίνηση στην ε, ε, χώρα και δεν σιωπούμε, εκφράσαμε ανησυχίες με αποφασιστικότητα και δημοσία και δημο, Νομίζω ότι εδώ έγκυται το πρόβλημα. Μέχρι τώρα τα ρωσικά δικαστήρια και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν έδειξαν να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα καθήκοντά τους και με ανεξαρτησία σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει δυσανάλογος αριθμός περιπτώσεων ρωσικών που φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικό εκπρόσωπο του ΙΕ για την εξαρτησία των δικαστών είπε μετά την πρόσφατη επίσκεψή τη στη Ρωσία ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για να εγγυάται την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος προστατεύοντας τους δικαστές από οποιαδήποτε μορφή πολιτικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεών τους. Αυτή είναι και η δική μας ε, άποψη. Τους επόμενες εβδομάδες και μήνες διάφορες ε, Δίκε κάτι, κ. βάλουν και άλλων και 12 δεδηλωτών Μποατνάγια θα ολοκληρωθούν οι δίκες. Αυτό ισχύει και για τη μεταθάνατον δίκη κατά του κυρίου Μαγνίσκη. Το ανώτατο δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση Χοντρακόσκη τον Αύγουστο. Εκφράσαμε σαφώς την άποψή μα για αυτές τις δίκες. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε λεπτομερώς τις δίκες στις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για στις 17 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις υποθέσεις εκ του σύνεγγυς. Το κράτος δικαίου θα πρέπει να είναι και είναι τομέας προτεραιοτήτων στην εταιρική μας σχέση για τον εξυγχρονισμό με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εφαρμόζουμε προγράμματα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και αυτός μας να βοηθούσε για να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί στη Ρωσία ένα σύστημα εφέσεων για ποινικά και αστικά, για ποινικέ και αστικέ υποθέσει. Και επίση και είπα θα συνεργαστούν με τη Ρωσία. Και για την εξαρτησία του δικαστικού τομέα. Πιστεύουμε ότι τέτοια προγράμματα έχουν δυνατότητα, δυνατότητα να παγιώσουν και να ενισχύσουν το νομικό περιβάλλον, βελτιώνοντα έτσι τι επενδύσει και το κοινωνικό κλίμα. Καλωσορίζουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε τη Ρωσία από αυτών των προγραμμάτων στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε να εκφράσουμε σαφώς ταυτόχρονα τις ανησυχίες μας. Και δημόσια όταν υπάρχουν προβλήματα. Και θα αναφερόμαστε και στη γενική κατάσταση όπως οι συγκεκριμένε υποθέσεις που αναφέρθηκαν στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Για να τελειώσει η συζήτηση να πω πως έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ε, ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει στο τέλος